15 μέρες ο κύριος Μπλουμ για να ε, προβάλλει ένσταση. Την Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 74 ε, του κανονισμού, θα υπογράψω 24 νομοθετήματα μαζί με το Συμβούλιο που εγκρίθηκαν στη συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία. Μαζί με τα σημερινά πρακτικά θα βρείτε και τις επικεφαλίδες όλων αυτών των αποφάσεων. Μέχρι